αρμόδια νομική επιτροπή που είναι η νομική επιτροπή. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες μου έδωσαν τον κατάλογο για τους διορισμούς στις διάφορες επιτροπές. Θα δημοσιευθούν στα πρακτικά και αν δεν διατυπωθούν ενστάσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα θεωρούν ως συγκεκριμένοι διορισμοί στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος και στην Υποεπιτροπή Άμυνας ο κύριος Σοφοκλής Σοφοκλέος. Και περνάμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση του κυρίου Μπέντσεν. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Ehm, er Ευχαριστώ. Πριν από 11 χρόνια οι Ισλαμικοί τρομοκράτε εξαπέλυσαν επίθεση κατά τι ιδέε της ελευθερίας στη Δύση. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής κίνησης επίθεσης που ήταν πάνω από 3.000. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν προβλέπετε στην ημερήσια διάταξη. Όμως δίκιο έχετε, καλό θα ήταν να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα θύματα της 11 ε, η Σεπτεμβρίου. Right. Πολύ ωραία.